και καθώς αυτό το έκανε βάσει πολύ συγκεκριμένων δικτών. Σας ευχαριστούμε για αυτή την ερώτηση. Θέλω να πω ότι ως προς τη διεύρυνση η Βόρεια Μακεδονία και η Αλβανία και επειδή αύριο θα είναι κρίσιμη ψηφοφορία ως προς το Σέγγεν εγώ θα ήθελα η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Κροατία να συμπεριληφθούν μόλις είναι έτοιμες και μόλις η Κροατία πληρεί όλες τις ε, τεχνικές προδιαγραφές. Ιδίως ό,τι αφορά το θέμα της επιστροφής των μεταναστών και των προσφύγων, προκειμένου να μην είναι παγιδευμένοι στα σύνορα μεταξύ Κροατίας και Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Ευχαριστούμε κύριος Μπορκία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ξεκίνησε μια διαδικασία αντεπροφούντης εξέτασης για την μελλοντική διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επειδή είναι πολλοί οι πολίτες της Αλβανίας που κάνουν αιτήσει ασύλου, αλλά και γιατί υπάρχει και το θέμα της απόρριψης της υποψηφιότητας της κυρίας Γκουλάρ. Εδώ βλέπουμε λοιπόν μια νέα τάση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση να διασπαθίζει τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων, ε, κάνοντα του δικού τη λογαριασμού και προβλέποντα ε, υποψηφιότητε για το μέλλον, λε και είναι η τέλεια λύση η Ευρωπαϊκή Ένωση για όλα τα προβλήματα. Η Αλβανία ε, είναι μέλος της, Ευρωπαϊκής, της Ισλαμικής Συμμαχίας και εδώ πολλά, πολλές σχολές που διδάσκουν το Κοράνι έχουν χρηματοδοτηθεί στην Αλβανία. Η Βόρεια Μακεδονία κάνει προπαγάνδα ότι πρέπει να φτάσει στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο στα Σκόπια. Πώ θα βλούμε λοιπόν την διεύρυνση ω μέτρο αναχέτηση τη ρωσική και κινέζικη εισβολή στα Δυτικά Βαλκάνια. Τι ακριβώ είναι η σωστή λύση που να ικανοποιεί όλου. Ευχαριστούμε ο κύριος Αλεξάνδροφ Γιορτάνοφ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Γαλλία δεν είναι κράτος που θα έκανα τέτοιου είδους φάλματα λόγω αμελίας. Είναι ένα κράτος που καταρχήν γνωρίζει τι κάνει. Όμως η απόφαση αυτή της Γαλλίας φαίνεται να εξυπηρετεί τα ρωσικά συμφέροντα στα Βαλκάνια. Και η Ρωσία, όπως γνωρίζουμε, είναι κατά της ευρωπαϊκής ανάπτυξης και της ευρωατλαντικής συνεργασίας ακόμη και στις ε, χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Η Ρωσία έχει ξεκινήσει και διεξάγει έναν, διεξάγει έναν υβριδικό ε, πόλεμο. Το σφάλμα αυτό του κυρίου Μακρό θα προκαλέσει προώρες εκλογές στη Βόρεια Μακεδονία και παρόλα αυτά δεν θα πρέπει να περιμένουμε εμείς την έκβαση των εκλογών, ούτε θα πρέπει να περιμένουμε τη σύνοδο στο Ζάγκρεμ. Διότι ο πρόεδρο Μακρό... Θα πει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τη νέα μακεδονική κυβέρνηση, βόρειο μακεδονική κυβέρνηση. Πράγμα που θα μας οδηγήσει σε μια πολιτική όξυνση. Ε, Εκτό ελέγχου. Θα έλεγα λοιπόν το Παρίσι να μην παίζει παιχνίδια με το Βελιγράδι και του υπόλοιπου. Ευχαριστούμε ο κύριο Μπενιφέη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι πεπισμένο ότι η πάυση των διαπραγματεύσεων που αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία ήταν ένα σοβαρότατο σφάλμα. Σήμερα βλέπουμε στι χώρε αυτέ να γίνεται σοβαρή δουλειά για την προσχώρησή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω δείχνουν η συμφωνία των Πρεσπών του 2018 μεταξύ Ελλάδα και Βόρεια Μακεδονία, καθώ και οι προσπάθειε που έκανε η Αλβανία πέρσι για να ευθυγραμμιστεί με τι προαπαιτήσει τη Ένωση. Η έναρξη των διαπραγματεύσεων θα ήταν σημαντικό για την έναρξη μια νέα περίοδου, γιατί θα έπρεπε να πάρουμε σοβαρά τα βήματα πρόοδου που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και να μην απογοητεύσουμε του νέου από τι χώρε αυτέ, αυτού του πολίτε που κοιτάζουν με εμπιστοσύνη αυτέ τι διαπραγματεύσει. Πολίτε που έρχονται από αυτέ τι χώρε και ε, έχουν φτιάξει τι οικογένειέ του και στη χώρα μου, την Ιταλία. Πρέπει σίγουρα να μεταρρυθμίσουμε το σύστημα τη Ένωση που δεν λειτουργεί καλά. Θα πρέπει να γίνει αυτό γιατί τα τελευταία χρόνια υπάρχει απέτηση για κάτι τέτοιο. Πρέπει να αλλάξει η λειτουργία των θεσμικών οργάνων, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει και πρόσχημα για να μπλοκάρουμε τα πάντα. Πρέπει να κάνουμε την Ευρώπη ισχυρότερη, συνεχίζοντα να ενώνοντα του λαού τη Επίρου μα. Ευχαριστώ πολύ. Mr. Ο κύριος Ντέλη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, ε, Πρόεδρε. Αξιότιμη κύριε Επίτροπε, αξιότιμη κυρία Υπουργέ. Την περασμένη εβδομάδα είδαμε τι συνέβη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και πού οδήγησε. Κατέστρεψε τελείως την αξιοπιστία της η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις μελλοντικές διευρύνσεις. Και τώρα δεν μπορούμε να απαιτούμε διάφορα πράγματα από τα κράτη της Δυτικής ε, Βαλκανικής, γιατί εμείς δεν ανταποκρινόμαστε στις υποχρεώσεις μας. Έχουν να κάνουν μεταρρυθμίσει. Οι διακρατικές σχέσεις ε, δεν είναι ο μονόδρομος. Καλό θα ήταν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ένωσης να καταλάβουν ότι αυτός που θίγεται ε, δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι προς όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενταχθούν τα κράτη αυτά. Υποτίθεται ότι θα πρέπει πρώτα να γίνει εσωτερική μεταρρύθμιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι άδικο όμως να ζητάμε από τα Δυτικά Βαλκάνια να περιμένουμε σταυρωμένα τα χέρια μέχρι να συμφωνήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να βρει λύση αποδεκτή από όλους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μίξερ για ένα λεπτό παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Η απόφαση του Συμβουλίου να μην αρχίσουν διαπραγματεύσεις με Βόρεια Μακεδονία και Αλβανία ήταν ιδιαίτερα λυπηρή και εκτό αυτού ήταν και τελείως λανθασμένη. Πολλά υπόθηκαν ε, σε σχέση με την αξιοπιστία μας, όχι μόνο σε αυτές τις δύο χώρες ε, που επιθυμούν να ενταχθούν στην Ένωση, αλλά και επέκεινα για όλη την περιοχή. Και είναι πραγματικά επέσχυντο το γεγονό ότι εσωτερικές πολιτικές ε, αιτίες οδήγησαν σε αυτό ε, δεν είναι ότι οι χώρε ε, που θέλουν να αρχίσουν διαπραγματεύσει δεν ήταν στο ύψο των περιστάσεων. Το αντίθετο. Ιδιαίτερα οι ηγέτε τη Βόρεια Μακεδονία επέδειξαν τεράστιο θάρρο και πήραν και πολύ μεγάλο πολιτικό κόστο για να λύσουν το θέμα με το γείτονά του ε, που εκκρεμούσε εδώ και χρόνια. Είναι κρίσιμο να διορθωθεί αυτό το σφάλμα πριν γίνει ανεπανόρθωτη ζημιά στην αξιοπιστία μας και στο κοινό συμφέρον για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Η κυρία Κοκαλάρη, για ένα λεπτό παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο Πρόεδρος Μακρό ήρθε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από δύο χρόνια περίπου στην Ολομέλεια και μας είπε τις απόψεις του για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Δημοκρατία είναι το καλύτερο σύστημα και ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθήσουμε το δρόμο της δημοκρατίας. Και συμφωνώ μαζί του, γι' αυτό θεωρώ αξιοθρύνητο αυτό το βέτο που άσκησε στην έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων ε, της Βόρειας Μακεδονίας και της Αλβανίας, γιατί κάτι τέτοιο διακυβεύει το σύνολο της διαδικασίας διεύρυνσης. Αυτή η διαδικασία διεύρυνσης ήταν πολύ χρήσιμο εργαλείο, ένας μηχανισμός για τις χώρες ε, και κίνητρο να προσπίσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και να ξεκινήσουν δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις. Θα πρέπει λοιπόν να ενθαρρύνουμε αυτές τις χώρες να εντείνουν τις προσπάθειές τους υπέρ της δημοκρατίας. Γιατί αν δεν είμαστε παρούσα η Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιοχή αυτή θα αφήσουμε το πεδίο ελεύθερο στην Τουρκία, στην Σαουδική Αραβία, στη Ρωσία και άλλες χώρες. Θα πρέπει η Ευρώπη να είναι ενωμένη και στα ανατολικά και στα δυτικά. Τώρα θα πρέπει να δράσουμε. Μάλιστα, ολοκληρώσαμε το κατάλογο των αγορητών και θα περάσουμε στη διαδικασία Catch the Eye. 13 Ομιλητέ ζήτησαν το λόγο στη διαδικασία αυτή, αλλά επειδή έχουμε μείνει λίγο πίσω στο χρονοδιάγραμμά μας, δεν θα μπορέσω να ικανοποιήσω όλους τους συναδέλφους που ζήτησαν το λόγο. Θα δώσω το λόγο μόνο σε έναν ανά πολιτική ομάδα, δίνοντας προτεραιότητα σε όσους δεν έχουν λάβει ακόμη το λόγο, ενώ ήταν παρόντες στην αίθουσα στη διάρκεια της συζήτησης. Ο κύριος Ποσπίσιλ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερο που η πλειοψηφία των συναδέλφων συμφώνησε ότι η απόφαση του Συμβουλίου ήταν εσφαλμένη. Έχουμε επανειλημμένως δηλώσει ότι είμαστε υπέρ της ένταξης των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οποιαδήποτε άλλη λύση θα ήταν εσφαλμένη. Μόνο θα αυξηθεί η επιρροή της Ρωσίας στην περιοχή αυτή, αν εμείς τους ε, στρέψουμε τα νότα και θα αποδυναμωθεί η δική μας παρουσία εκεί. Ε, με τι πρόσωπο θα μιλήσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους αν τους κλείνουμε την πόρτα. Νομίζω ότι είναι προ όφελο και προ το συμφέρον τη Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσει με τι χώρε αυτέ και στους ε, συναδέλφου που έχουν αμφιβολίες για το κατά πόσο είναι σκόπιμο κάτι τέτοιο, σα διαβεβαιώ ότι μιλούμε για έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Αυτό δεν σημαίνει προσχώρηση. Οι ενταξιακέ διαπραγματεύσει είναι χρονοβόρε. μπορούν να κρατήσουν χρόνια ολόκληρα, αλλά δίνουμε την ελπίδα και την ευκαιρία στι χώρε αυτέ κάποια μέρα να γίνουν μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πραγματικά η απόφαση του κ. Μακρόν είναι κατά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Uh, thank you. Κυρία Ward, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε ως φίλη των Δυτικών Βαλκανίων. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι και η Αλβανία και η Βόρεια Μακεδονία κάποια στιγμή θα γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όντως, πραγματοποίησα σημαντικά και επιτυχή βήματα στην ενταξιακή τους πορεία και πραγματικά αυτή η κοινή προσπάθεια της Γαλλίας και της ε, Ολλανδίας και της Δανίας να σαμποτάνε αυτή την προσπάθεια ήταν αξιοθρή, αξιοθρύνητη. Μάλιστα, η Βόρεια Μακεδονία και η Αλβανία ε, προηγούνται κάποιων κρατών μελών. Και οι δύο χώρε, για παράδειγμα, έχουν κυρώσει τη συνθήκη τη Κωνσταντινούπολη. Ενώ η δική μου πατρίδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, ακόμη δεν έχει κάνει κάτι τέτοιο. Ενώ η Βουλγαρία αργεί και χρονοτριβεί. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε έγκριση για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων στο μέλλον, γιατί θα επηρεαστεί η εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολο των Δυτικών Βαλκανίων, αν δεν επιδείξουμε πολιτική ακεραιότητα και άνοιγμα. Είμαι πεπισμένη ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το μέλλον της Ευρώπης έγκυται στην ενότητα με τα Δυτικά Βαλκάνια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Αουστρεβίτσιους. Πρόεδρε, Επίτροπε, συνάδελφοι. Για μια Ευρώπη ενιαία σε ειρήνη και αναπτυσσόμενη. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία γειτονία και προσχώρηση για να επιτρέψουμε στι γειτονικέ χώρε να δημιουργήσουν ε, οικονομία τη αγορά και να έχουν μορφωμένου και καταρτισμένου πολίτε. Επίση, πρέπει να προωθήσουμε την περιφερειακή συνεργασία και σταθερότητα. Τα προγράμματα δράση και συμφωνίε εταιρική σχέση ε, προβάλλουν αυστηρά κριτήρια για του γειτονέ μα και πρέπει να τα ικανοποιήσουν. Όμω, ξεχνάμε λίγο να τηρήσουμε εμεί τι δικέ μα υποσχέσει. Αυτό δεν είναι σωστό. Οι υποψήφιε χώρε μπορεί να μην είναι πανέτοιμε για να προσχωρήσουν σήμερα, όμω πρέπει να κοιτάξουμε τι, συμβαίνει, τι θα συμβεί στο απότερο μέλλον. Πρέπει να ε, εξισορροπήσουμε προσπάθειε ε, όπω αυτέ τη Ρωσία, που με τι απόπειρέ του ε, κάνουν προτάσει για κοντόφθαλμα πολιτικά παιχνίδια, ενώ η προοπτική διεύνηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει το καλύτερο, την καλύτερη προοπτική για το βιωτικό επίπεδο, την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αν δεν το πράξουμε αυτό θα πρέπει ε, να δούμε πώς ε, αυτή η θεώρηση για την, ε, κοινή, για την προσχώρηση είναι σημαντική. Ευχαριστώ πολύ και αγαπητοί συνάδελφοι. Αυτό που είδαμε στην τελευταία σύνοδο κορυφή είναι πραγματικά ιστορικό σφάλμα για την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία να παραμένουν κλειστέ οι θύρε. Δεν είναι απλώ προσβολή για τι κυβερνήσει του, αλλά για τη νέα γενιά κυρίω. Είναι ένα μοιραίο μήνυμα που στέλνουμε σε όλη την περιοχή. Στο παρελθόν, γενναίε ολόκληρε στα Βαλκάνια μεγάλωναν χωρί ε, ε, προοπτικέ για πραγματική πρόοδο. Αυτό του οδήγησε να φύγουν, να ψάξουν να βρουν την τύχη τους αλλού. Ε, όλοι πόνταραν για, την επόμενη γενιά ε, ότι θα είχε μια πραγματική ευκαιρία να παραμείνει στη χώρα της. Ε, τώρα με αυτή την απόφαση ε, να μην ανοίξουν οι διαπραγματεύσεις παρά το γεγονός ότι έχουν πληρώσει όλα τα κριτήρια, παγώνουν ε, οι ελπίδες. Οι άλλοι, κάποιοι άλλοι δεν θα περιμένουν πολύ να καλύψουν αυτό το κενό που αφώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδιαίτερα Ρωσία, Τουρκία, Κίνα, Κατάρ, ακόμα και Σαουδική Αραβία διαγωνίζονται για να υπάρξει πολιτική συνεργασία στην περιοχή. Αυτό μάλλον δεν είναι προς το δικό μας συμφέρον. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λεμπρετών.

Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που το Συμβούλιο μπλόκαρε τις διαπραγματεύσεις ένταξης Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Αλβανία είναι πασίδλο ε, μια χώρα όπου ενδυμεί η διαφθορά και ασφικτιά η κοινωνία. Ο ένας στους τρεις νέους είναι άνεργος, σύμφωνα με τα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας. Βέβαια υπάρχει μια μεταρρύθμιση στη δικαιοσύνη εδώ και χρόνια με πάρα πολύ ανισχυτικά αποτελέσματα. Μια ε, επιτροπή ανεξάρτητη με διεθνού εμπειρογνώμονε έχει ε, βγάλει τους ε, διεφθαρμένους ε, δικαστές, ε, από τους 17 έχουν μείνει ε, δύο στο ανώτατο δικαστήριο και στο συνταγματικό από εννέα, ένας μόνο. Ε, ας μην γελιόμαστε. Δεν ε, αρμόζει στην Αλβανία να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 28 έκτου του 2019 έλεγε η βελγική εφημερίδα Λεσουάρ ότι είναι ναρκοκράτος υπό την επίρρεια των διακινητών. Ο κύριος Παπαδημούλης. Κύριε Πρόεδρε, σε λίγες ώρες η ολομέλεια του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου θα ψηφίσει με συντριπτική εκτιμώ πλειοψηφία ένα ψήφισμα όλων σχεδόν των πολιτικών ομάδων το οποίο ζητά από το συμβούλιο να διορθώσει άμεσα αυτό το ιστορικό λάθος. χαιρετίζουμε την ιστορική συμφωνία των πρεσπών και στέλνουμε ένα μήνυμα εμείς από το ευρωκοινοβούλιο στους λαούς της βόρειας μακεδονίας και της αλβανίας ότι η ευρωπαϊκή ένωση δεν είναι ούτε ανέντιμη ούτε αναξιόπιστη. και στέλνουμε και ένα μήνυμα στον πρόεδρο εμμανουέλ μακρόν ότι το όχι του που πρέπει να το διορθώσει γρήγορα δεν παίζει το παιχνίδι της σταθερότητας και της δημοκρατίας ούτε υπηρετεί τα ευρωπαϊκά συμφέροντα υπηρετεί τα συμφέροντα των εθνικιστών του ερντογάν του πούτιν και της αστάθειας και στην ευρώπη και στα βαλκάνια. γι' αυτό τον χειροκροτούν και οι ακροδεξιοί μέσα στην αίθουσα. Έχω σημειώσει το αίτημα υποβολή ερώτηση με την μπλε κάρτα, αλλά επειδή έχουμε μείνει πολύ πίσω ε, και είμαστε και στη διαδικασία του Κασδιά. θα απορρίψω το αίτημα για ερώτηση με μπλε κάρτα. Λυπάμαι. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Επίτροπο Χάν εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους παρόντες ειλικρινά για την συντριπτική υποστήριξη της αξιόπιστης διαδικασίας ε, προσχώρησης για τις δύο χώρες, Βόρεια Μακεδονία και Αλβανία πρέπει να δοθεί το πράσινο φως, να μπορέσουμε να αρχίσουμε τις ε, προενταξιακές διαπραγματεύσεις. Να αρχίσουμε, δεν λέμε ότι θα μπουν αύριο ή μεθαύριο. Ε, μιλούμε για διαπραγματεύσεις. Είναι μια πολυετής διαδικασία αυτή. Χρόνια ολόκληρα ε, χρειάζεται για να χτίσεις αξιοπιστία και αρκούν λίγα λεπτά ή λίγες ώρες για να την κρεμίσεις την αξιοπιστία αυτή. Και μέχρι κάποιο βαθμό συνέβη στα Δυτικά Βαλκάνια και όχι μόνο πρέπει να σας πω, όχι μόνο στα Δυτικά Βαλκάνια. Με την απόφαση αυτή ως Ευρωπαϊκή Ένωση χάσαμε πολλή αξιοπιστία, ε, πολλή εμπιστοσύνη που μας χαρακτηρίζει και διεθνώς και παγκοσμίως. Και αυτό το λέω και σε σχέση με τα όσα συμβαίνουν στην άμεση γειτονία μα. Υπάρχει μια σειρά προβλημάτων που αναδύονται. Κοιτάξτε τι γίνεται στο Λίβανο. Για να μην μιλήσω για τη Μέση Ανατολή γενικότερα. Την Ισία, η πολιτική κατάσταση εκεί. Ιδιαίτερα έφραυση. Αλγερία. Συγκεχημένη η πολιτική κατάσταση. Και δεν μπορώ παρά να ελπίζω ότι εκείνοι που ευθύνονται για την τωρινή κατάσταση δεν είχαν επίγνωση του τι σημαίνει για το κύρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό παγκοσμίω και ιδιαίτερα στη γειτονία μας. Και τι σημαίνει για τις δυνατότητες που έχουμε επιρροής, επίλυσης ε, προβλημάτων και επιβολής ακόμα. Και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανακτηθούν αυτά. Επειδή εγώ είμαι φύση αισιόδοξο. Βλέπω το ποτήρι μισό γεμάτο. είναι να πιστεύω ότι θα διορθωθούν τα πράγματα. Και μάλιστα μπορώ να ακούσω και τα διάφορα επιχειρήματα που ακούστηκαν τους τελευταίους μήνες. Γιατί να μην αρχίσουν ήδη από τώρα οι διαπραγματεύσεις. Και τα λαμβάνω σοβαρά υπόψη. Αλλά καμιά φορά έχω την αίσθηση ότι τα επιχειρήματα αυτά που προβάλλονται είναι προφάσεις. Για να μην πούμε ρητά και κατηγορηματικά ότι κοιτάξτε με αντίθετο με τη διεύρυνση. Πάντω, ένα από τα επιχειρήματα που ακούσαμε από τη Γαλλία και από κάποιε άλλε χώρε ήταν ότι πριν την επόμενη διεύρυνση χρειάζεται εμβάθυνση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βελτίωση ε, της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, συνεργασίας κλπ. Προσωπικά σας λέω ότι Συμφωνώ. Τα κατανοώ όλα αυτά πάρα πολύ. Αλλά δεν κατανοώ καθόλου για ποιο λόγο αυτά τα δύο πρέπει να γίνουν διαδοχικά. Υπάρχει κάλλιστα η δυνατότητα και έχει και νόημα και ρεαλιστικό είναι και ό,τι θέλετε να γίνουν παράλληλα αυτές οι διαδικασίες. Γιατί χρόνια θα χρειαστούν και οι δύο. Ε, τώρα όμως, εάν αρχίσουμε να συζητάμε την εμβάθυνση πρώτα και μετά σε ένα απότερο χρόνο τις ε, μελλοντικές ε, διευρύνσεις, τότε αυτές οι χώρες έχουν μια προοπτική διεύρυνση στη δεκαετία του 2030. Ε, δεν νομίζω να θεωρείται προοπτική η ένταξη σε αυτό. Ε, και μπορώ να σας διαβεβαίωσω κυρίες και κύριοι ότι οι υπηρεσίες μου και εγώ προσωπικά και θεωρώ και εκείνος που θα με αντικαταστήσει, εκείνη που θα με αντικαταστήσει, θα κάνουν ό,τι μπορούν για να ε, κοιτάξουμε ε, την μέθοδο της διαδικασίας προσχώρησης, ουδής δεν είναι τέλειος, αλλά και παντού, χωρούν και πάντα βελτιώσεις. Πολλά από όσα άκουσα ισχύουν ήδη. Ε, το κράτος δικαίου, η δυνατότητα των διαπραγματεύσεων, και η διαπραγμάτευση δεν σημαίνει αυτόματα ένταξη. Είναι μια διαδικασία. Λοιπόν, αυτό θα κάνουμε και ελπίζω ε, να ε, υπάρξει και η αντίστοιχη προσήλωση και ενθουσιασμός. Και επιτρέψτε μου να σας πω μια μικρή ιστορία, πιο σύντομη από ό,τι ακούγεται. Το 2013 που ήμουν επίτροπο για την περιφερειακή πολιτική στι Βρυξέλλε, έκανα ε, ένα μικρό σεμινάριο με εκπροσώπου τη κοινωνία των πολιτών από τη Βόρεια Ιρλανδία. Που τότε μου έδειξαν τα διάφορα προγράμματα που είχαν τα έργα για την ε, συμφιλίωση στη Βόρεια Ιρλανδία ε, και πώς τα προωθούσαν και πώς τα οργάνωναν. Και δεν μπορώ παρά να σας πω ότι το 90% των συμμετεχόντων το 2013 ήταν εκπρόσωποι κρατών από την πρώην Ιουκοσλαβία. Και ήξεραν πάρα πολύ καλά γιατί συμμετείχαν εκεί σε αυτά τα προγράμματα. Γιατί ξέρουν απολύτως ότι η ειρήνη, η σταθερότητα και η ευημερία στα Δυτικά Βαλκάνια μπορούν να έρθουν μόνο εφόσον υπάρχει ένταξη σε ένα γενικότερο σύνολο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ και πάλι για αυτό το ηχηρό μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξία. Αυτό θα εκπέμψουμε και θέλω να απευθυνθώ στον πρόεδρο της Βόρειο-Μακεδονικής Βουλής και να του ευχηθώ καλή επιτυχία και να τον ευχαριστήσω ιδιαίτερα προσωπικά για τις πολλές πρωτοβουλίες που ανέλαβε τους τελευταίους μήνες έτσι ώστε η χώρα να ε, ανοίξει για την Ευρώπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Τουπουράινεν, εκ μέρους του Συμβουλίου. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της ε, Βουλής της Βορείου Μακεδονίας, αξιότιμη Ευρωβουλευτέ, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συζήτηση αυτή και επ' να ευχαριστήσω και τον Επίτροπο Χάν για την ε, διαρκή προσήλωσή του στη διαδικασία της διεύρυνσης. Η συζήτηση αυτή με έχει πείσει ακόμη περισσότερο ότι η στήριξή μας στα Δυτικά Βαλκάνια, η υποστήριξη εκεί της ε, ευρωπαϊκής προοπτικής είναι στεναρή και μόνιμη. Και υπό το φως των δηλώσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα επανέλθουμε στο θέμα το, της διαβίωσης προς τα Δυτικά Βαλκάνια πριν τη Σύνοδο Κορυφή στο Ζάγκρεπ τον Μάιο του 2020 που σημαίνει ότι θα συνεχιστεί το έργο, δεν θα πρέπει να εγκαταλείψουμε που δεν είναι. Επίσης θα ήθελα να σας ε, υπενθυμίσω ότι η συμφωνία για την έναρξη των διαπραγματεύσεων, των ενταξιακών διαπραγματεύσεων είναι μόλις το πρώτο βήμα μιας ε, μακράς διαδικασίας. Και εγώ ένιωσα απογοήτευση και προσωπικά αλλά δεν νομίζω ότι είναι τώρα σκόπιμο να κολλήσουμε σε αυτά που συνέβησαν την περασμένη εβδομάδα και παρόλο που να μπαίνουμε σε αυτό, μπορούμε να πούμε σε αυτόν τον πειρασμό, καλό θα ήταν να μην δακτυλοδεικνύουμε ούτε να ξεβροστιάζουμε και να ονομάζουμε κάποιον. Θα πρέπει να περάσουμε στο μέλλον, στα επόμενα βήματα και προσεκτικά να σχεδιάσουμε τα επόμενα βήματα για να σημειώσουμε επιτυχία σε μια διαδικασία που ούτω ή άλλω θα είναι μακρά και χρονοβόρα και θα απαιτήσει σκληρή και εργόδη προσπάθεια από όλου. Πάντω, κάνουμε ένα προσεκτικό και διεξοδικό απολογισμό τη κατάσταση και θα προχωρήσουμε στη συνέχεια. Πάντως θα ήθελα να κρατήσω την αισιοδοξία και την ελπίδα μου. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να είμαι και ρεαλίστρια σε ό,τι αφορά την προοπτική για τους επόμενους μήνες. Σέβομαι πλήρως το έργο που υλοποίησαν και οι δύο χώρες, η Βόρεια Μακεδονία και η Ελβανία, και τι μέχρι τώρα προσπάθειές του. και θα ήθελα να ενθαρρύνω και τις δύο χώρες να συνεχίσουν στο ίδιο πνεύμα και να υλοποιήσουν τις μεταρρυθμίσει που ξεκίνησαν ε, για χάρη και προς το συμφέρον των πολιτών τους, γιατί ό,τι είναι καλό για εκείνου είναι και θα είναι θετικό και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ για τη συζήτηση και για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ. Έχω λάβει 7 σχέδια ψηφίσματος για τη συζήτηση, μετά τη συζήτηση αυτή και προέρχονται από το ID, το ECR, τους Πράσινους, την QNGL, τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, την ομάδα Renew Europe και το ELK. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την συμμετοχή σας στη συζήτηση αυτή, να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Χάν, την κυρία Τουπουράινεν, τον ε, πρόεδρο της Βορειομακεδονικής Βουλής που ήταν ε, παρόν στη συζήτηση και να κηρύξω το πέρας της συζήτησης αυτού του σημείου. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης που προβλέπει δήλωση της είπα της ε, εκπροσώπου για την εξωτερική πολιτική και αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα την κατάσταση στο Ιράκ και ιδιαίτερα τη βίαιη καταστολή των διαμαρτυριών των νέων και των φοιτητών στο Ιράκ. Πριν κηρύξω την έναρξη της συζήτησης, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι για, το, για τη διαδικασία ερωτήσεων με μπλε κάρτα και για το Catch the Eye θα έχετε τη δυνατότητα να ε, εγγραφείτε και ηλεκτρονικά στον κατάλογο. Οπότε να έχετε μαζί σας τον, ε, την κάρτα ψηφοφορία σας για την συζήτηση με την μπλε κάρτα. Μπορείτε να το δηλώσετε από τώρα, δεν χρειάζεται να περιμένετε το, τέρας, το πέρας της συζήτησης. Και μια και έχουμε μείνει λίγο πίσω, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι δεν θα είμαι σε θέση να δώσω το λόγο στη διαδικασία του Κατσδιάη σε όλους τους ομιλητές ενδεχομένω. Τη συζήτηση θα την ξεκινήσει η κυρία Τουπουράινεν που θα μας παρουσιάσει τη θέση του εκ μέρους ε, της ΥΠΑΤΣ εκπροσώπου για την εξωτερική πολιτική και Αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε να έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι βουλευτέ. Στι αρχέ Οκτωβρίου, οι διαμαρτυρίε που ξεκίνησαν στη Βαγδάτη και μετά που εξαπλώθηκαν στι υπόλοιπε πόλει του Ιράκ οδήγησαν σε κλιμάκωση και σε ε, συγκρούσει ε, και εκατοντάδε θανάτου, με τουλάχιστον 600 τραυματίε. Το διαδίκτυο, 6.000 ε, ε, τραυματίες τουλάχιστον. Εδώ τα τηλεοπτικά δίκτυα καλύπτουν την ε, επίθεση σε άοπλους διαδηλωτές και η Ευρωπαϊκή Ένωση το έκανε τελείως σαφές από τις 3 Οκτωβρίου ότι ελπίζουμε οι δυνάμεις καταστολής να δείξουν εγκράτεια στη χρήση βίας και συγκράτηση και να φροντίσουν να μην υπάρξουν άλλες βίες επιθέσεις. Μετά τις δηλώσεις των, ε, των, αρχών, των, ε, είπα, των αρχών του Ιράκ πρέπει να προστατευθεί η ελευθερία έκφρασης και του ε, διαδηλώνει όλων των πολιτών του Ιράκ καθώς και η ελευθερία του τύπου θα πρέπει να μην αντιμετωπίζεται με καταστολή κάθε έκφραση των Ιρακινών. Οι διαμαρτυρίες φαίνεται ότι ξεκίνησαν αυθορμήτως από νέους που ζήτησαν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, καλύτερες ευκαιρίες και να δοθεί τέρμα στο καθεστώς διαφθοράς. Οι προσδοκίες τους και τα παράπονά τους είναι νόμιμα και θεμητά και δεν θα πρέπει να υποτιμούνται. Οι νέοι σε όλη τη Μέση Ανατολή ε, βγαίνουν στους δρόμους ακριβώς με τα ίδια αιτήματα παντού. Ε, ταυτόχρονα οι προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει το Ιράκ είναι ιδιαίτερες. Η χώρα επιτέλους βγαίνει από μια περίοδο μακράς, μακρών εχθροπραξιών, πρέπει να περάσει σε φάση ανοικοδόμησης, αλλά πρέπει να καλύψει και τις προσδοκίες των πολιτών για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες για όλους. Αυτές οι προσδοκίες θα πρέπει να εκπληρωθούν εφόσον θέλουμε το Ιράκ να σταθεροποιηθεί μακροπρόθεσμα οι αξιόπιστες και αποτελεσματικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις δεν μπορούν να αναβάλλονται. Θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η διαφθορά καταλήλως. Αυτό ε, είναι αποφασιστικό για, τον, για να χτιστεί μια ανθεκτική χώρα με ισχυρούς δημοκρατικούς θεσμούς και ισχυρό δημοκρατικό πολίτευμα. Η τωρινή κυβέρνηση του Ιράκ έχει προτείνει μια φιλόδοξη ατζέντα μεταρρυθμίσεων που θα πρέπει να υλοποιηθεί κατεπηγόντως. Η ύπατη εκπρόσωπο, πήγε στη Βαγδάτη το καλοκαίρι και ήδη από τότε πρόσφερε την υποστήριξή τη στην ατζέντα μεταρρυθμίσεων τη κυβέρνηση, με επικέντρωση την προσφορά και την προμήθεια υπηρεσιών στον πληθυσμό τη χώρα. Τα τελευταία χρόνια πάντοτε βρεθήκαμε στο πλευρό των Ιρακινών και τη δουλειά του για ανοικοδόμηση και συμφιλίωση τη χώρα. Στις αρχές του 2018 συν, ε, διοργανώσαμε μια διεθνή διάσκεψη για την ανοικοδόμηση του Ιράκ και Τώρα ε, προσπαθούμε να τηρήσουμε τις υποσχέσεις που είχαμε αναλάβει στην συνδιάσκεψη. 300 ε, εκατομμύρια ε, εκταμιεύτηκαν τα τελευταία δύο χρόνια για να στηρίξουμε τις μεταρρυθμίσεις και να υπάρξει βιώσιμη δημιουργία θέσεων αναπασχόλησης, κυρίως για τις νέες γενιές τους νέους που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή των πρόσφατων διαμαρτυριών και διαδηλώσεων. Τα τελευταία χρόνια έχουμε κοιτάξει να αποναρκοθετήσουμε τα πανεπιστήμια και τα νοσοκομεία της χώρας, προκειμένου να έχουν όλη πρόσβαση εκεί και προσπαθήσαμε να οργανώσουμε την Εθνική Συμφιλίωση συνεργασία με τις κυβερνητικές αρχές, καθώς και με τις διοκτικές αρχές, τις αρχές ασφάλειας της χώρας να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον ασφαλές και κυρίως εκείνοι οι ίδιοι να συμμορφώνονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις απαιτήσει για τις βασικές ελευθερίες. Δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι το Ιράκ έχει ε, καταφέρει σημαντική πρόοδο τα τελευταία δύο χρόνια μετά την εδαφική ήττα του Νταές στις γενικές εκλογές του 2018 που ε, ε, οδήγησαν σε μια ειρηνική μεταφορά της εξουσίας προς τη νέα κυβέρνηση και τις τοπικές κυβερνήσεις. Εμείς οι Ευρωπαίοι ανέκαθεν λέγαμε ότι θέλουμε ο λαός του Ιράκ να ε, καταφέρει και να κερδίσει την ειρήνη, του, την ειρήνη που του αξίζει. Αυτό ζητάει τώρα ο λαός της χώρας. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να είμαστε στο πλευρό τους και να ε, στηρίζουμε τους πολίτες του Ιράκ για μια πιο συμμετοχική, ολοκληρωμένη και σταθερή δημοκρατία. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα ακολουθούν οι ομιλητές εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων. Αλλά προηγουμένως θα ήθελα να σας παρακαλέσω να τηρείτε το χρόνο σας γιατί έχουμε κάποια καθυστέρηση. Για 1,5 λεπτό παρακαλώ το λόγο έχει ο κύριος Κίρτσος από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Έχουμε μια κρίση μεταξύ Ιράν και Σαουδικής Αραβίας ταραχές στο Λίβανο, εισβολή στη Συρία και άλλες εξελίξεις που τονίζουν τη σημασία ενός σταθερού Ιράκ σε μια περιοχή εύθραυστη και δύσκολη. Η οικονομία του Ιράκ μετά από 20 χρόνια πόλεμο ανακάμπτει και με χρόνια παρουσία του λεγόμενου Ισλαμικού κράτους στην επικράτειά του. Το δυναμικό της χώρας είναι τεράστιο το Ιράκ είναι ήδη ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός του ΟΠΕΠ, 4,6 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. 3,5% ανάπτυξη ε, ε, προβλέπουν οι οικονομολόγοι και 4% το 2020. Θα πρέπει να ζητήσουμε από την κυβέρνηση να αξιοποιήσει το οικονομικό δυναμικό της χώρας για να αντιμετωπίσει τα μελήματα και τις ανησυχίες των πολιτών που οδήγησαν στις πρόσφατες κοινωνικές ε, αναταραχές. Έχει χάσει τον έλεγχο της κατάστασης και των δυνάμεων ασφαλείας η κυβέρνηση θα πρέπει εμείς να μιλήσουμε υπέρ της ε, εφαρμογής του προγράμματος 13 σημείων για μεταρρυθμίσεις που έχει ε, εξαγγείλει η κυβέρνηση και να γίνει μια ανεξάρτητη διερεύνηση ε, του θανάτου πάνω από 100 διαδηλωτών. Ευχαριστώ πολύ. Για δύο λεπτά. Το λόγο έχει η κυρία Πύρη, εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, το, τους μήνες αυτούς δεκάδες χιλιάδες ε, κατέβηκαν στους δρόμους ε, σε περιοχές ε, με πλειοψηφία σιτών. Ήταν άοπλοι οι διαδηλωτέ και σε καμία περίπτωση δεν ήταν κίνδυνο για την ασφάλεια. Και παρόλα αυτά ήταν στιγμή η καταστολή από τι δυνάμει ασφαλεία. Τουλάχιστον 110 έχασαν τη ζωή του. Χιλιάδε τραυματίστηκαν και σύρθηκαν στι φυλακέ. Και μάλιστα ένα παραστρατητικό ακροβολιστή ε, σκότωσε πολλούς στους δρόμους της Βαγδάτης. Είναι απαράδεκτες αυτές οι παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα πρέπει να τις τηλητεύσουμε κατηγορηματικά και ρητά. Επίσης να προστατεύσουμε του διαδηλωτέ. τους ε, Οι διαμαρτυρίες κρατούν μήνε. Οι περισσότεροι είναι άνεργοι γιατί δεν υπάρχουν στοιχειώδεις βασικές υπηρεσίες. Εδημεί η διαφθορά η καταστολή συνεχίζεται και οι δράσεις της κυβέρνησης ε, είναι προβληματικές, ε, προκαλούν ανησυχία. Δεν ε, υπάρχει καμία αλλαγή. Το αντίθετο μάλιστα. 25 Οκτωβρίου είναι η προθεσμία της κυβέρνησης να προσαγάγει στη δικαιοσύνη τους αυτούργους της δολοφονίας άοπλων πολιτών. Δεν μπορούμε να δίνουμε βίαιη απάντηση σε εύλογες απαιτήσει του λαού. Θα πρέπει να έχουμε ε, κοινωνικές ε, μεταρρυθμίσεις και ε, πάταξη της διαφθοράς. Κάτι τέτοιο απαιτεί πολιτικό θάρρος. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στέκεται στο πλευρό των Ιρακινών και είναι πρόθυμο να βοηθήσει τις αρχές αν θέλουν πραγματικά να επενδύσουν χωρίς αποκλεισμού στις οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις της χώρας. Είμαστε έτοιμοι να αποδείξουμε ότι είμαστε δίκαιος ε, και αξιόπιστος εταίρος της περιοχής αυτής. Ευχαριστώ. Η κυρία Αλσαχλάνη, εκ μέρους του Ρινιού για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω στα Σουηδικά, αλλά θα ήθελα πρώτα να απευθύνω έναν ε, χαιρετισμό προς την Ιρακινό λαό στα Αραβικά. 110 ε, άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε λίγες μέρες, χιλιάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν, ε, πυροβολήθηκαν στο κεφάλι, στο στήθος από ακροβολιστές που πυροβολούσαν για να τους σκοτώσουν, ενώ ήταν άμαχοι, ήταν πολίτες που σήκωναν την ε, Ιρακινή σημαία διεκδικώντας τα δικαιώματά τους, το τέλος της διαφθοράς, το δικαίωμά τους στην απασχόληση, το δικαίωμά τους στην παιδεία, διεκδικούσαν μια αξιοπρεπή ζωή οι Ιρακινοί, οι νέοι που διαδήλωναν στο Ιράκ. Διαδήλωναν γιατί ζητούσαν μία πατρίδα που θα τους προστατεύει. Δυστυχώς η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργό αποφάσισε ε, να διεξαγάγει μια έρευνα, αλλά διαπιστώνουμε ότι σε όλη τη χώρα καταπατάται το Σύνταγμα. Θα πρέπει να παταχθεί επιτέλους η διαφθορά που είναι ενδημική στη χώρα. Δεν υπάρχει ούτε ένας υπουργός, που να αναλαμβάνει την ευθύνη για τους θανάτους αυτούς ε, άμαχων πολιτών. Κανένας ε, δεν κατηγορήθηκε ως αυτούργός ε, για την εντολή της βίαιης αυτής καταστολής των διαδηλωτών. Ποιος έδωσε την εντολή για τέτοια άσκηση βίας ε, είχαμε την ανατροπή του Σαντάμ Χουσέιν, μετά την άφηξη των Αμερικανών και μετά την, τον ΤΑΕΣ, μετά τον ΤΑΕΣ είχαμε την Αλκάιδα, ο Ιρακινός λαός ανέκαθεν έδινε μάχη για την αξιοπρέπειά του και στο Ιράκ και στην Ευρώπη. Οφείλουμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση να απαιτήσουμε αλλαγή της κατάστασης και να επιμείνουμε σε αυτό. Λυπάμαι που έχουμε μόνο συζήτηση χωρίς ψήφισμα. Πάντως θα πρέπει να επιμείνουμε για να αφογκραστεί η κυβέρνηση τα αιτήματα των διαδηλωτών. Θα πρέπει ο Ιρακινός λαός να γίνει σεβαστός και να μπορέσει να ζήσει μέσα σε αξιοπρέπεια. Νόημα από τους πράσινους. Συνάδελφοι, είναι δικαίωμα των ανθρώπων στο Ιράκ να βγαίνουν στο δρόμο και να διαμαρτύρονται. Όμως εκατοντάδες έχουν τραυματιστεί, μάλλον έχουν θανατωθεί, 400, τουλάχιστον έχουν ε, τραυματιστεί και είναι πολλοί δημοσιογράφοι που έχουν φυλακιστεί. Είναι σαφές αυτό που λένε οι οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι, δυνάμεις, οι δυνάμει του Ιράκ επιτίθενται σε άοπλους πολίτε και ε, υπάρχουν έρευνες για... δεν υπάρχουν μάλλον ακόμα έρευνες για τους αυτούργους και τους δράστες. Ε, αντιθέτως, ναι, περισσότεροι διαμαρτυρητές φυλακίζονται και καταστέλλονται οι διαδηλώσεις. Αυτό λοιπόν ανησυχεί εμά και το κοινοβούλιο ολόκληρο. Εδώ και δύο χρόνια υπάρχει μια εξεταστική αποστολή τη ε, Ευρωπαϊκή Ένωση που συνεργάζεται με το Υπουργείο του Ιράκ. Πρέπει να κοιτάξουμε τι γίνεται με το τομέα ασφαλεία στο Ιράκ και πρέπει τουλάχιστον να δούμε πόσοι, 95 ε, τουλάχιστον έχουν ε, κρατηθεί και φυλακιστεί και να δούμε γιατί είναι τόσο βία η καταστολή των διαδηλώσεων τις τελευταίες εβδομάδες. Θα πρέπει κυρία Τουπουράινεν να μας πείτε τι συνέπειες έχει συναγάγει η αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ιράκ, τι έρευνες θα υπάρξουν για τους δράστες και τους αυτοργούς και πώς θα φροντίσουμε να σταθεροποιηθεί η περιοχή χωρίς να υπάρχουν και άλλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τις επιθέσεις αυτές και πώς θα φροντίσουν για αυτό τα Υπουργεία του Ιράκ και οι αρχέ τη χώρα. Συνάδελφοι, επιτέλου στην Ολομέλεια πρέπει να μιλήσουμε και για τι δικέ μα αποστολέ στο εξωτερικό. Thank you, Mr. Mariani, one minute. Ο κύριος Μαγιανή, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το Ιράκ είναι ε, ε, μια χώρα πληγωμένη ε, από το 2003, από την Αμερικανική επέμβαση, ε, από τις φρικαλαιότητες στην Ινεβή, στον Μπαρ, στα Σαλαχεντίν ε, του Ισλαμικού κράτους. Επανειλημμένα έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματα και κυριαρχία από Αμερική και Τουρκία. 5.200 είναι Αμερικανοί στο Ιράκ και αυτούς που έβγαλε ο Τραμπ από τη Συρία τους πήγε εκεί. Το 2018 το ΝΑΤΟ υποτίθεται ότι θα έκανε αποστολές εδραίωσης της εξουσίας. Από τον, τον Οκτώβριο ε, υπάρχει στο Ταρμπίν ένα προσκύνημα που έρχονται ε, κατά εκατομμύρια οι και έχουμε διαδηλώσεις. Οι θρησκευτικοί ηγέτες ζητούν ε, από την κυβέρνηση να ανταποκριθεί στα αιτήματα της κοινωνίας και των διαδηλωτών. Καλά κάνουμε και μιλάμε για αυτές τις διαδηλώσεις και την καταστολή που καταδικάζουμε. Αλλά εμείς το 2003 ε, μπήκαμε εκεί πέρα χωρίς να σκεφτούμε το μέλλον και χωρίς την ε, νεολαία να σκεφτούμε γιατί καταστρέψαμε τη χώρα. Το Ιράκ είναι κατεστραμμένο και εμεί φέρνουμε μεγάλο τμήμα της ευθύνης γι' αυτό. Ένα λεπτό, κυρία Φωτίγκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπήρξε μια περίοδος ελπίδας στο Ιράκ μετά ε, την ε, ήττα του ISIS, παρά τις δυσκολίες. Και τώρα βλέπουμε μαζικές διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς, κατά της ανεργίας με κακές δημόσιες υπηρεσίες και η αντίδραση της κυβέρνησης ήταν ε, μάλλον υπερβολική και οδήγησε σε πολλούς θανάτους. Και μάλιστα ε, υπήρχαν και ίχνη ε, προβοκάτσιας και με ακροβολιστές ελεύθεροι σκοπευτές πυροβολούν τους διατηρητές και όλο και πιο πολλοί νέοι σκοτώνονται, δολοφονούνται και πάνω από 6.000 είναι οι τραυματίες. Θα πρέπει οπωσδήποτε να υποστηρίξουμε την κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Αβδέλα Μαχτή, αλλά θα πρέπει επίσης να ζητήσουμε ε, να αναλυφθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να ε, προσαχθούν στη δικαιοσύνη Η υπετη των παραβιάσεων ε, της καταστολής. Ο Πρόεδρος. Υπάρχει γαλάζια κάρτα, αλλά πραγματικά τώρα ε, οι ομιλητές μιλούν εξ ονόματος των πολιτικών τους ομάδων. Η κυρία Φωτίγκα μίλησε εξ ονόματος του ECR, οπότε δεν μπορώ να δεχτώ γαλάζια κάρτα. Για ένα λεπτό το λόγο έχει η κυρία Ντέιλι από την GUE NGL, εξ ονόματος της ομάδας της. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σαν σήμερα πέρσι ήμασταν στο Ιράκ και πριν από τρεις εβδομάδες ο νεαρός που μας είχε ξεναγήσει πυροβολήθηκε και φίλοι του που επίσης έπαιρναν μέρος στις διαδηλώσεις ε, έχασαν τη ζωή τους. Αυτό που πιο πολύ μας, μας στεναχωρεί είναι ότι στην Ιρλανδία οι Ιρακινοί φίλοι του λένε ότι κανείς δεν φαίνεται να νοιάζεται στον κόσμο. Εκατοντάδες έχουν δολοφονηθεί, εκατοντάδες έχουν τραυματιστεί και δεν υπάρχει ούτε ένα πρωτοσέλιδο. Είναι πραγματικά παράδεκτο αυτό για τον αποκατισμό αυτή τη χώρα. Οι άνθρωποι αυτοί θέλουν απλά πράγματα, νερό, ηλεκτρισμό, δουλειέ και δεν του τα δίνουν. Γιατί, Γιατί είναι το κληροδότημα της παράνομης εισβολής των ΗΠΑ που πήραν τα ε, περιουσιακά στοιχεία του Ιράκ, έκλεψαν, έκλεψαν τους φυσικούς χώρους και καταλήστεψαν τη χώρα αφήνοντας ένα καθεστώς διαφθοράς. Είναι χρεωμένη για πάντα η χώρα αυτή και πραγματικά θα πρέπει η τωρινή κυβέρνηση ε, που είναι υπέρ των ΗΠΑ να ε, είναι τελείω διαφορετική. Εδώ δεν μπορούμε να είμαστε ταυτόχρονα λίγο φιλικοί προ τη Συρία, λίγο φιλικοί προ το Ιράκ και να μην βρίσκουμε ποιοι είναι υπεύθυνοι για του πυροβολισμού. Εγώ δεν ξέρω, δεν πιστεύω ότι είναι ξένοι πράκτορε που δρούν σε αυτή την περιοχή απλώ. Ευχαριστούμε για του μη εγγεγραμμένου από ο μη εγγεγραμμένο κ. Καστάλντο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι διαδηλώσει ε, των τελευταίων εβδομάδων ε, στο Ιράκ έχουν να κάνουν με νέου νέους ε, και Κούρδους και από το Ιράκ για τι βασικέ υπηρεσίε που δεν προσφέρονται στο Ιράκ. Χρειάζεται μια πλήρη αναθεώρηση του πολιτικού συστήματο. Η απάντηση των αρχών ήταν βία, παράδεκτη και φρικαλέα. Εκατοντάδε έχασαν τη ζωή του λόγω τη συμπεριφορά των διοκτικών αρχών. Αυτή η βία καταστολή των διαδηλώσεων είναι απαράδεκτη και συνάδελφοι θα πρέπει να απευθύνουμε έκκληση στην Ιρανική κυβέρνηση για να σεβαστεί τι βασικέ ελευθερίε του λαού θα πρέπει να εγγυηθούμε την προστασία των πολιτών. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στου πολίτε που εργάζονται για του λίγου και όχι για του πολλού να δρουν ανενόχλητοι στην Συρία, στη Λιβύη, στο Σουδάν, σε οποιαδήποτε τέτοια χώρα που δημιουργούν αυτή την ε, παγκόσμια στάθεια. Είναι μια από τι πολλέ χώρε όπου έχουν επιβληθεί αντιδημοκρατικά μέτρα με την καταστολή των μέσων μαζική ενημέρωση και την ε, πλήρη ανεξέλεγκτη δράση των δημόσιων αρχών. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να δούμε πώ εντείνονται οι εντάσει εντό και εκτό των χωρών χωρών, μοντέλα ανάπτυξη που δεν βασίζονται στην κοινωνική συμμετοχή όλων. Και μόνο αν επιτρέψουμε σε όλου να εκφραστούν ελεύθερα θα μπορέσουμε να βρούμε τι κατάλληλε λύσει. Ο κύριο Ρουί Δεβέσα, εκ μέρου των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το Ιράκ, γνωρίζουμε όλοι, δεν είναι μόνο το λίκνο του πολιτισμού μας, αλλά ταυτόχρονα είναι και από τα ελάχιστα δημοκρατικά σχέδια φιλελεύθερου τύπου, τουλάχιστον απόπειρα ε, δημοκρατικού σχεδίου φιλελεύθερου τύπου στη Μέση Ανατολή. Και ω τέτοιο χρήζει αμέριστη πολιτική, διπλωματική, ακόμη και οικονομική υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τούτου λεχθέντο, είναι προφανέ ότι οι εξελίξει τη τελευταία εβδομάδα ε, είναι απαράδεκτες και θα πρέπει να τις καταδικάσουμε. Θα πρέπει να πετήσουμε απονομή ευθυνών. Θα πρέπει να διελευκανθούν η άνω των 150 θάνατοι ε, με ε, πυροβολισμούς κατά αόπλων διαδηλωτών που απλώς διαμαρτύρονταν διεκδικώντας βελτιώσεις οικονομικές και κοινωνικές στο Ιράκ. Θα πρέπει λοιπόν να επιβεβαιώσουμε τη συμπαράστασή μας στον Ιρακινό λαό υπέρ της ευημερίας του και υπέρ της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράκ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σμπαουθά Δίαθ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω στα Ισπανικά. Και θα ήθελα να απευθυνθώ στην κυρία Μογκερίνη φυσικά που είναι η αρμόδια. Εδώ και ένα χρόνο το Ιράκ βρίσκεται εγκλωβισμένο σε ένα κύκλο βίας, δυσαρέσκειας και ματέωσης. Θα πρέπει να αντιστρέψουμε αυτή τη στάση με τη βοήθειά μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Χιλιάδες Ιρακινοί νέοι κατέβηκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν κατά της διαφθοράς, κατά της έλλειψης στοιχειωδών υπηρεσιών και κατά της ανεργίας. Αυτά τα ακούσαμε και από τους συναδέλφους. Είναι εύλογες οι απαιτήσει που όμως αντιμετωπίστηκαν με εκφοβισμό των δημοσιογράφων, περιορισμό του ίντερνετ και χρήση στιγνής βίας εκ μέρους της κυβέρνησης. Γι' αυτό θα πρέπει να στελιτεύσουμε και να καταδικάσουμε αυτή την αδικαιολόγητη χρήση βίας που μέχρι στιγμής στήχησε τη ζωή σε πάνω από 150 διαδηλωτές και άφησε ε, χιλιάδες τραυματίες. Τα θύματα βέβαια θα πρέπει να αποζημιωθούν και οι ευθύνες των δραστών θα πρέπει να αποδοθούν. Αυτός ο κύκλος της δυσαρέσκειας και της βίας θα συνεχιστεί όσο συνεχίζονται τα βασικά προβλήματα διακυβέρνησης που έχει το Ιράκ και που γνωρίζουμε όλοι ποια είναι. Η διαφθορά, η πελατοκρατία και ένα πολιτικό σύστημα που επιδεινώνει το, το διαχωρισμό της χώρας, το διχασμό. Επίσης θα πρέπει να απαιτήσουμε από την κυβέρνηση του Ιράκ την τήρηση των διεθνών υποχρεώσεών της, ε, να τεθεί ένα τέρμα στη βία και να εγγυηθεί τα δικαιώματα της ελευθερίας έκφρασης, της ελευθεροτυπίας και της ελευθερίας του ε, συνέρχεσθε των Ιρακινών πολιτών. Αυτή είναι υποχρέωση και καθήκον μας και αυτές θα πρέπει να είναι οι απαιτήσει μας απέναντι στην Ιρακινή κυβέρνηση. Ευχαριστώ. Η κυρία Τοβαλιέρη, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στη Βαγδάτη και σε άλλες πόλεις του Ιράκ έχει ξεκινήσει μια βία η καταστολή φοιτητών και νέων ανέργων που διαδηλώνουν εδώ και εβδομάδες κατά της διαφθοράς και της ε, ε, μιζέριας, της φτώχειας που εξαπλώνεται. Οι νέοι είναι το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. 4 στους 10 είναι χωρίς δουλειά και χωρίς μέλλον. Οι ειδικέ δυνάμεις πυροβολούν ανοιχτά κατά των διαδηλωτών, προκαλώντας θανάτους, τραυματισμούς και αυθαίρετες συλλήψεις. Εδώ ε, ο ιστός της, της ο πολιτικός ιστός είναι διεφθαρμένος. Ε, και υπάρχει ε, ουσιαστικά πόλεμος κατά των ίδιων των πολιτών με το πρόσχημα ότι πολεμούν την τρομοκρατία. Και υπάρχει και καταστολή των χριστιανών και των γυναικών. Στην επικράτεια του Ιράκ, στο, το ISIS ε, σκοτώνει και θανατώνει συστηματικά τους ε, χριστιανούς και επιβάλλει στις γυναίκες την κάλυψη με μαντήλα. Εδώ θα πρέπει να προασπιστούμε τις αρχές μας και να αποφύγουμε την μαζική ε, μετανάστευση από αυτές τις χώρες ε, που καταπιέζονται οι διάφορες κοινότητες του πληθυσμού. Ευχαριστούμε, κύριος Μπορένα Άρθα. Πρόεδρε, από την αρχή του ε, Οκτωβρίου διαδηλώνουν στο Ιράκ νέοι και ζητούν καλύτερη ζωή, καλύτερες υπηρεσίες και όχι διαφθορά. Και τους πατάσουν με πυροβολισμούς με αντλίες ε, νερού. Ε, έχουμε εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες. Θα πρέπει να σταματήσουν αυτά. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ζητήσουμε από την κυβέρνηση της Βαγδάτης να ακούσει ε, το λαό της και να χαλιναγωγήσει τις δυνάμεις ασφαλείας. Θέλουν να μιλούν ελεύθερα και να χρησιμοποιούν ελεύθερα το ίντερνετ οι νέοι. Η Ιρακινή κυβέρνηση ε, οφείλει να προστατεύει το δικαίωμα του συνεταιρίζει, του συνέρχεστε της ελευθερίας του λόγου βάσει των διεθνών υποχρεώσεων. Ανησυχούμε επίσης για τα συλλογικά αστυνομικά μέτρα ε, κατά των πολιτών που έχουν συγγενείς που υποτίθεται ε, νίκουν στο Ισλαμικό κράτος. Αυτό θα οδηγήσει σε νέο κύμα βίας ε, στο Ιράκ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπαρτόλο, ε, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρο. Στη Βαγδάτη και στι γειτονικέ περιοχέ είναι εκατοντάδε οι νεκροί και χιλιάδε οι τραυματίε στο πλαίσιο τη τη βία που έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο και διατρέχει ολόκληρη τη χώρα εδώ και εβδομάδε. Αυτά τα φαινόμενα βία δεν ξεκινάνε από το πουθενά, αλλά έχουν να κάνουν με την κοινωνία και την οικονομία προβλήματα σοβαρότατα που μαστίζουν μια χώρα που εδώ και χρόνια προσπαθεί να ξεφύγει ένα πόλεμο που τη γονάτισε. Αυτή η δυσφορία έχει φέρει εκατοντάδε χιλιάδε νέου φοιτητέ και πολίτε, κανονικού πολίτε, στι ε, πλατείε και τις, ε, τους δρόμους των απόλυων του Ιράκ για να πάυσει η ε, διαφθορά που είναι πανταχού παρούσα και εμποδίζει την ανάπτυξη τον εξυγχρονισμό τη χώρα. Το ποσοστό τη ανεργία των νέων είναι πραγματικά πρόβλημα με την αύξηση του κόστου ζωή και την έλλειψη βασικών υπηρεσιών που οδηγούν σε μια νέα κοινωνικού χαρακτήρα σύγκρουση. Εδώ λοιπόν πρέπει να επιτρέψουμε το δικαίωμα του διαδηλών ε, με τρόπο ειρηνικών και η κυριακή κυβέρνηση να επιτρέψει την ελευθερία τη έκφραση, δρώντα με σεβασμό ε, το ίδιο και οι δυνάμει ασφαλεία τη χώρα για να σεβαστού, γίνουν σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταγγείλει κάθε μορφή βία και να φροντίσει να επαγρυπνεί για τέτοιε εξελίξει και στο μέλλον. Πρέπει να εγγυηθούμε τη τη χώρα αυτής σε πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο για την ίδια τη χώρα, το Ιράκ και την ευρύτερη περιοχή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. our list. Μάλιστα, ολοκληρώσαμε τον κατάλογο των ομιλητών. Περνάμε στη διαδικασία του Catch the Eye. Ο κύριος Τσιχοντάρου. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οφείλω να ομολογήσω ότι είμαι τρομοκρατημένος αλλά και εμβρόντιτος γιατί δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι στον 21ο αιώνα θα είμαστε μάρτυρες ε, τέτοιας στιγμής χρήσης βίας. Ε, είμαι γιατρός ε, και είδα σε νοσοκομεία θύματα τέτοιας βίας κατά νύμπορων πολιτών. Μόνο ένα σατανικό μυαλό θα μπορούσε να επινοήσει κάτι τέτοιο. Είμαι πραγματικά τρομοκρατημένος γιατί η ελευθερία έκφρασης που είναι θεμελιώδης δικαίωμα όλων των πολιτών καταστρατηγείται οικειοθελώς τον 21ο αιώνα. Και αυτό εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί τέτοια κατάσταση έχουμε σε πολλά μέρη του κόσμου. Ίσως θα πρέπει να καθίσουμε όλοι σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων και να επινοήσουμε ένα σχέδιο για να αντιμετωπίσουμε τέτοιε καταστάσει, ώστε τέτοιε φρικαλαιότητε να μην επαναληφθούν στο μέλλον. Επαναλαμβάνω, είμαι τρομοκρατημένο, αγανακτισμένο, εξοργισμένο και σα απευθύνω έκκληση να βρούμε μία λύση από κοινού για να αποτρέψουμε επανάληψη τέτοιων φαινομένων στο μέλλον. Η κυρία Κόνετσνα. Σα ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, τα πορίσματα της Εξεταστικής Επιτροπής του Ιράκ είναι σαφή. Ε, ο θάνατος 157 ατόμων στις πρόσφατες διαδηλώσεις οφείλονται στην ε, βαναυσότητα των ε, δυνάμεων ασφαλείας. Η καταστολή που άσκησαν ήταν στιγμή. Οι δυνάμεις ασφαλείας έπρεπε να προστατεύσουν τους διαδηλωτές, όχι να τους σκοτώνουν. Αυτό δείχνει ότι η δημοκρατία βρίσκεται σε κίνδυνο. Ελπίζαμε να είναι σε καλύτερη κατάσταση το Ιράκ. Αν όμως η απάντηση στους διαδηλωτές είναι ε, πυροβόλα, όπλα και κανόνια νερού, αυτό δείχνει η παναχώρηση της δημοκρατίας στο Ιράκ. Η βαναυσότητα των δυνάμεων ασφαλεία θα πρέπει να στυλιτεύεται όπου και αν λαμβάνει η χώρα, ακόμη και στην Καταλωνία. Είναι πραγματικά ντροπή να γινόμαστε μάρτυρες τέτοιων καταστάσεων. Η κυρία Βόρτ. Πρόεδρε, χιλιάδες διαδηλωτές, κυρίως νέοι, διαδηλώνουν σε όλο το Ιράκ κατά της διαφθοράς και κατά της ενεργείας. Απαιτούν μια κυβέρνηση που θα λογοδοτεί και καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες τους καταστέλει όμως, ε, τους καταστέλουν οι αρχές, ε, διοκτικές αρχές της χώρας, οι αρχές ασφαλείας, οι οποίες έχουν τραυματίσει χιλιάδες και θανατώσει εκατοντάδες. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει ανεξάρτητη έρευνα για αυτούς τους φόνους και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι αρχές πρέπει αμέσως να απελευθερώσουν όλους τους διαδηλωτές, οι οποίοι ε, δεν, είχαν, δεν κατηγορήθηκαν με κάτι το αξιόμεμπτο και κάτι που πραγματικά συνέβη. Απλώς άσκησαν το δικαίωμα δικαίωμά του για να διαδηλώσουν, να συμμετέχουν σε μια διαδήλωση και να επικρίνουν την κυβέρνηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι εγκληματίε. Ε, και επίση δεν μπορεί να υπάρχει τέτοια επίθεση κατά των διαδηλωτών και φήμωση ενώ προσπαθούν να εκφραστούν. Η κυβέρνηση του Ιράκ είναι υποχρεωμένη βάσει του διεθνού δικαίου να προστατεύει το δικαίωμα ελεύθερη έκφραση, του διαδηλώνων και τη ε, ελεύθερη ε, έκφραση. Ευχαριστούμε ε, το Ιράκ είναι μια χώρα κατεστραμμένη. Δεν μα εκπλήσει που διαδηλώνει ο κόσμο και διαμαρτύρεται. Ούτε μα εκπλήσει που η κυβέρνηση είναι άχρηστη. Η ζημιά που έχει γίνει στη χώρα αυτή, το Ιράκ, έχουμε δει τίποτα τόσο χάλια τα τελευταία 30 χρόνια. Είναι απίστευτο και πραγματικά είναι λυπηρό γιατί τα ευρωπαϊκά κράτη δεν είναι αθώα. Βεβαίω όλα αυτά τα ξεκίνησαν οι Αμερικάνοι και φταίνε. Βεβαίω ήταν το θέμα των πόρων και το να αλλάξει το καθεστώ για να. Αλλά η φτώχεια και η εγκατάλειψη, αυτό έχει βλάψει τον ίδιο τον λαό. Είναι χιλιάδες αυτοί που έχουν ε, πεθάνει μέχρι τώρα. Αυτός ο αριθμός των τωρινών θανάτων είναι μικρός σε σχέση με ε, το, το παρελθόν. Οι βουλευτές δεν νοιάζονται να κάνουν κάτι για το λαό. Νοιάζονται πιο πολύ για τα όπλα. Ε, εδώ λοιπόν φαίνεται να είναι πολύ δύσκολο οι δυτικέ δυνάμεις να βοηθήσουν μια χώρα χωρίς να την ε, καταλυστέψουν και να την ε, παραβιάσουν όλα τα δικαιώματα. Εδώ ολοκληρώνεται ο κατάλογο του ΚΑΣΕ. Α, θα δώσω το λόγο στην κυρία Τουπουρά. Είναι να μιλήσει εξ ονόματο τη Αντιπροέδρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υπάτη εκπροσώπου τη Ένωση για θέματα εξωτερική πολιτική και ασφαλεία. Έχετε το λόγο. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, Επιτρέψτε μου να πω ότι ήταν πολύ χρήσιμη αυτή η ανταλλαγή απόψεων και φυσικά πάρα πολύ επίκαιρη. Επ' ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω τους βουλευτές για τις παρεμβάσεις, τα σχόλια και τις προτάσεις τους.